Ε, κύριε Διαμεσολαβητά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ευρωβουλευτές, ε, δικηγόροι, εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Καλώ ήρθατε στην Επιτροπή Ελέγχου του Προπολογισμού. Ζητώ συγγνώμη ξανά του κυρίου Στά, ε, πρώτο αντιπροέδρου τη Επιτροπή μα. Η ε, ακρόαση αυτή ενεγράφει στην ημερήσια διάταξη μετά από πρόταση της ηγήτριας συναδέλφου κυρίας Γκρέσλε, στην οποία θα δώσω σε λίγο το λόγο. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω κύριε Διαμεσολαβητά ε, που δεχθήκατε την πρότασή μας. Ε, σας έχουμε ανάγκη, χρειαζόμαστε τα φώτα σας ε, και τις γνώσεις που έχετε από την υψηλή σας θέση για τη συνεργασία των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων με τους ε, πολίτες. Περιμένουμε με ανυπομονησία και με προσοχή θα ακούσουμε την άποψή σας για όλα τα θέματα κοινοποίησης, ε, διοικητικής δυσλειτουργίας και καταγγελίες ε, ε, σχετικά με την προστασία των ε, υπαλλήλων και τις πειθαρχικέ διαδικασίες, όλα αυτά τα θέματα που ενδιαφέρουν και απασχολούν την κυρία Γκρέσλε. Θα ήθελα να καλωσορίσω και το δικηγόρο κύριο Ζάνο Νοέλ Λουί. Καλωσορίσατε εξοχότατε. Μας ενδιαφέρει πάρα πολύ και το θέμα της προστασίας των προσώπων αλλά και τις καταγγελίες και κοινοποίησης διαφόρων λειτουργιών που αντιμετωπίζουμε στη λειτουργία των θεσμικών μας οργάνων. Τέλος θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Κάρεν Βίλιαμς, η οποία θα λάβει και είναι το λόγο. Είναι αρμόδια για την υπηρεσία ερευνών και επιθαρχικών κυρώσεων της Γενικής Διεύθυνσης Ανθρωπίνων Πόρων και θα ήταν ενδιαφέρον να ακούσουμε την άποψή σας κυρία Διευθύντρια. Χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση θα δώσω το λόγο στην εισηγήτριά μας, την κυρία Ίγκε Γκρέσλε. Ah oui, euh, donc elle, conclura, elle conclura. Α, θα κλείσει κυρία Γκρέσλε, δεν θα κάνει την εισαγωγή, τα συμπεράσματα. Ωραία. Ε, κύριε Δημοσιολογητά, παρακαλώ, έχετε το λόγο. Euh, Ευχαριστώ πολύ, κύριε Οντή, για την πρόσκληση αυτή και για την θερμή σας υποδοχή. Χαίρομαι ιδιαίτερα που βρίσκομαι εδώ στην Κοκομπή, στην Επιτροπή σας και θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω την κυρία Γκρέσλε διότι με κάλεσε να σας πω τις απόψεις μου για το θέμα αυτό του whistleblowing που πολύ γρήγορα ε, μεταφράζεται, πολύ δύσκολα μεταφράζεται στα γαλλικά και σε σχέση με τις πειθαρχικές κυρώσεις. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Επιτροπή Ελέγχου του Προπολογισμού για την πρόσκληση που μου απίθυνε για να μιλήσω εδώ πέρα σήμερα για πιθανές ελλείψεις ε, στους κανόνες περί καταγγελίας λειτουργιών και τις πειθαρχικές διαδικασίες. Όπως ενημέρωσα ήδη την ε, κυρία Γκρέσλε, οι παρατηρήσεις μου θα αναφερθούν όχι μόνο στον κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης, αλλά και στους ε, κανόνες που διέπουν τον αυτή την υπηρεσία κατά πολέμησης απάτης. Είχα λοιπόν δύο ερωτήματα κατά νου όταν προετοίμαζα αυτές τι παρατήσεις. Το πρώτο είναι πώς μπορούμε να προωθήσουμε καλύτερα την ηθική συμπεριφορά και να αποθαρρύνουμε την ανήθικη συμπεριφορά των υπαλλήλων και αυτή θα είναι η σκοπιά υπό την οποία θα δω τα πράγματα. Δεύτερον είναι ποια είναι η σωστή κατανομή ευθυνών μεταξύ Όλαφ και υψηλόβαθμων στελεχών στους διάφορους ε, φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα παραμείνω λοιπόν στο πλαίσιο αυτής της, ε, του θεσμικού διαχωρισμού των αρμοδιοτήτων. Να σας πω επίσης πως σήμερα δεν θα κάνω λεπτομερείς ε, προτάσεις. Θα κάνω μια αναγνώριση των ε, προβλημάτων και του στόχου που θα πρέπει να επιτύχουν οι μεταρρυθμίσεις κατά την άποψή μου. Όμως αυτή τη στιγμή είναι πρόωρο να προτείνουμε συγκεκριμένες διατυπώσεις για αλλαγή των νομικών διατάξεων. Θα ήθελα επίσης να ξεκαθαρίσω ευθύς εξ αρχής πως οι παρατηρήσεις μου δεν έχουν ε, στόχο να αποτελέσουν συνολική πρόταση για τις απαραίτητες αλλαγές είτε στον κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης είτε στο νομικό πλαίσιο λειτουργίας του Όλαφ. Θα ήθελα όμως να ξεκινήσω με το να θέσω ένα βασικό ζήτημα που αφορά τη λειτουργία του Όλαφ. Ο Όλαφ συστάθηκε πριν από 12 χρόνια μετά την πτώση της Επιτροπής Σαντέρ. Και τις παρατηρήσεις μιας Επιτροπής Ανεξαρτήτων Ειδικών ε, για τις περιπτώσεις απάτης ε, και νεποτισμού στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο κανονισμός 1073 του 99, ο λεγόμενος κανονισμός Όλαφ, δίνει αρμοδιότητες στον Όλαφ να κάνει εξωτερικές έρευνες μέσω επιτοπίων επιθεωρήσεων και ελέγχων στα κράτη-μέλη. Ο κανονισμός επίσης προβλέπει πως ο Όλαφ μπορεί να κάνει εσωτερικές έρευνες εντός των θεσμικών οργάνων, γραφείων και αποκεντρωμένων υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή η εσωτερική πτυχή είναι αυτή η οποία μας απασχολεί σήμερα. Είναι λοιπόν σημαντικό να ξεκαθαρίσουμε πως οι αρμοδιότητες του Όλαφ για εσωτερικές έρευνες δεν βασίζονται αποκλειστικά στον κανονισμό του. Ο κανονισμός ο ίδιος απαιτεί κάθε θεσμικό όργανο να λάβει μια απόφαση η οποία θα προβλέπει εσωτερικές έρευνες από τον Όλαφ υπόδειγμα απόφασης περιέχεται στην ε, διοργανική συμφωνία μεταξύ Συμβουλίου, Κοινοβουλίου και Κομισιών που υιοθετήθηκε ταυτόχρονα με τον κανονισμό. Το υπόδειγμα απόφασης προβλέπει πως ο Όλαφ ε, μπορεί να διερευνεί πιθανές περιπτώσεις όχι μόνο απάτης, διαφθοράς και άλλων ε, ανάλογων δραστηριοτήτων, αλλά και συμπεριφοράς η οποία θα μπορούσε να καταλήξει σε πειθαρχικές διαδικασίες. Βεβαίω, ε, όπω ε, καταλάβατε, δεν είναι αυτή η ακριβή διατύπωση. Θα σα διαβάσω τώρα. Στοιχεία τα οποία οδηγούν σε υποψίες ε, ύπαρξης απάτης, διαφθοράς ή άλλη παράνομη δραστηριότητα η οποία βλάπτει τα συμφέροντα τη κοινότητα ή η κατάσταση η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει σε απαλλαγή από τα καθήκοντα στην περίπτωση στην οποία κάποιο δεν συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις του ως υπάλληλο και μπορεί να οδηγήσει σε πειθαρχικές ή ποινικέ διώξεις ή μη ε, συμμόρφωση με τις ε, υποχρεώσεις των ε, υπαλλήλων που δεν περιέχονται στον οργανισμό υπηρεσιακής κατάστασης. Όλο αυτό είναι μία περίοδος το 2004 είχαμε έναν απλούστερο ορισμό που μπήκε στο άρθρο 86 κανονισμού υπηρεσιακή κατάστασης και πλέον το άρθρο αυτό επιτρέπει στην αρχή διορισμού ή στον Όλαφ να ξεκινήσει μια διοικητική έρευνα εάν υποπέσει στην αντίληψή τους κάποιο στοιχείο οποιασδήποτε παράληψης ε, υπαλλήλου ή πρώην υπαλλήλου να συμμορφωθεί ε, είτε μέσω είτε μέσω παράληψης με τα όσα ισχύουν. Υπάρχει λοιπόν εδώ πέρα μια διπλή ασάφεια όσον αφορά τον ρόλο του Όλαφ. Και θα την εξηγήσω παρά το ότι μας ενδιαφέρει μόνο η δεύτερη ασάφεια αυτή τη στιγμή. Η πρώτη ασάφεια είναι το ότι ο Όλαφ ονομάζεται Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης, αλλά ο κανονισμός του δίνει ένα πολύ ευρύτερο ρόλο προστασίας των ε, κοινωτικών συμφερόντων από παρατυπίες, κάτι το οποίο δεν σημαίνει οπωσδήποτε κάποια κακοήθεια. Δεύτερη, ε, η δεύτερη ασάφεια είναι η δυνατότητα που του δίνεται να ερευνήσει πιθανές τέτοιες πράξεις, ακόμα και αν δεν υπάρχει βλάβη των οικονομικών σφαιρών της κοινότητας. Κατά την άποψή μου είναι ιδιαίτερα σημαντική και προκαλεί βλάβη η δεύτερη ασάφεια, γιατί μπορεί να δημιουργήσει σύγχυση για το τι μπορεί και τι θα έπρεπε να κάνει ο Όλαφ. Επίσης θεωρώ πως υπονομεύει αυτό το οποίο κατά την άποψή μου θα έπρεπε να είναι η ευθύνη της διοίκησης ε, των θεσμικών οργάνων για να διασφαλιστεί η ηθική συμπεριφορά. Θα μπω σε λεπτομέρειες αργότερα, αλλά πριν ε, γίνει αυτό θα ήθελα να κάνουμε εισαγωγή στο θέμα της παροχής πληροφοριών. Παρά το ότι δεν χρησιμοποιείται η λέξη καταγγελία, στα άρθρα 22α και 22β ε, γενικώ θεωρείται πως αναφέρονται σε αυτή την περίπτωση. Κατά βάση τα άρθρα αυτά κάνουν δύο πράγματα. Πρώτα απ' όλα ορίζουν τις συνθήκες υπό τις οποίες κάποια είδη καταγγελίας προστατεύονται από αντίπεινα από πλευράς ε, των θεσμικών οργάνων και αυτό βέβαια είναι κάτι το πολύ σημαντικό και ενδιαφέρει τα μέλη της Επιτροπής σας όμως δεν είναι το αντικείμενο της σημερινής μου ομιλίας. Το δεύτερον που υπάρχει σε αυτές τις ε, διατάξεις και εδώ πέρα αναφέρομαι στο άρθρο 22α είναι ότι επιβάλλει υποχρέωση στους υπαλλήλου να καταγγείλουν. Συγκεκριμένα το άρθρο 22α υποχρεώνει τους υπαλλήλους να αναφέρουν πιθανές περιπτώσεις απάτης, διαφθοράς, λοιπόν παρανόμων δραστηριοτήτων ή επαγγελματικής συμπεριφοράς η οποία θα μπορούσε να αποτελεί μη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις των υπαλλήλων. Κατά βάση, ένας υπάλληλο πρέπει να συμμορφωθεί είτε ενημερώνοντας την ιεραρχία του, είτε πηγαίνοντας απευθείας στον Όλαφ. Στην πρώτη περίπτωση, τα άτομα τα οποία ενημερώνονται πρέπει να μεταδώσουν άμεσα τις πληροφορίες αυτές στον Όλαφ. Οι διατάξεις αυτές λοιπόν μας οδηγούν σε κάποιες παρατηρήσεις. Πρώτα απ' όλα, το πεδίο εφαρμογή είναι αβέβαιο γιατί δεν είναι σαφές πώς σχετίζονται με μια άλλη διάταξη το άρθρο 21α. Το άρθρο αυτό αφορά τις περιπτώσεις στις οποίες ένας υπάλληλος λαμβάνει διαταγές, τις οποίες θεωρεί παράτυπες, ή μπορεί να δημιουργήσουν σοβαρές ε, δυσκολίες. Δεν ορίζονται αυτές οι πιθανές καταστάσεις, αλλά φαίνεται πιθανόν πως ζητήματα ηθικής θα ε, προκύψουν εδώ πέρα, τουλάχιστον σε κάποιες περιπτώσεις. Δεύτερον, η διατάξει περί καταγγελίας δεν ε, θέτουν το βάρο ε, τη ευθύνη στην διοίκηση των ε, εν λόγω θεσμικών οργάνων για να δράσει προληπτικά. Η μόνη δράση η οποία απεφαίνεται να προβλέπεται είναι να απευθυνθούν στον Όλαφ εάν η εν λόγω συμπεριφορά θεωρείται σοβαρή. Θεωρώ πως δεν είναι ικανοποιητική αυτή η προσέγγιση είτε στην πράξη είτε και επί της αρχής. Στην πράξη οι ασάφειες οι οποίες ανέφερα για τον ρόλο του Όλαφ φαίνεται πως δεν έχουν επιληθεί μέσω της εμπειρίας σύν χρόνο. Δεν είναι σαφέ, τουλάχιστον για μένα, το εάν ο Όλαφ θεωρεί ότι τα καθήκοντά του συμπεριλαμβάνουν τι εσωτερικέ έρευνε στην περίπτωση πιθανή συμπεριφορά που δεν επηρεάζει τα οικονομικά συμφέροντα τη κοινότητα. Υπάρχει λοιπόν αυτή τη στιγμή μια ε, σύγχυση η οποία θα μπορούσε να προκύψει όχι μόνο μεταξύ καταγγελόντων και ε, ανθρώπων οι οποίοι θα ήθελαν να κάνουν καταγγελίες αλλά και της διοίκηση των θεσμικών οργάνων και πιθανώς και του ιδίου του Όλαφ. Ο κίνδυνος αυτός αυξάνεται ε, αν δούμε την περίπλοκη διατύπωση του άρθρου 22α του κανονισμού υπηρεσιακής ε, κατάστασης, η οποία αντιγράφει την κακή διατύπωση του υποδείγματος απόφασης που σας ανέφερα πριν. Επιπλέον, επί της αρχής, το καθήκον του να προάγεται η ηθική συμπεριφορά ε, εντός ε, των θεσμικών οργάνων θα έπρεπε να είναι αρμοδεότητα της φυσικής ηγεσία και της διοίκησης το να λέμε πως αυτό αφορά αρμοδιότητα κάποιου άλλου δεν τους ενθαρρύνει να προωθήσουν μια τέτοια συμπεριφορά. Αυτά τα οποία είπα μέχρι στιγμή ε, αφορούν τα προβλήματα τα οποία βλέπω στο εφιστάμενο νομικό πλαίσιο. Στο υπόλοιπο μέρο τη ε, παρουσίασή μου θα εξετάσω του στόχου, του οποίου θεωρώ πω θα πρέπει να έχει κατά νου ο κοινοτικό νομοθέτη όταν προχωρήσει αναθεώρηση αυτού του νομικού πλαισίου. Πρώτο και κύριο, ο κανονισμό υπηρεσιακή κατάσταση θα πρέπει να εκφράσει σαφώ το ότι τα θεσμικά όργανα και ειδικά η διοίκηση είναι υπεύθυνοι για την διατήρηση της ηθικής συμπεριφοράς και την πρόληψη μη, και την πρόληψη μη συμπεριφοράς. Θα πρέπει λοιπόν να ενθαρρυνθεί και να διευκολυνθεί η καταγγελία αντιεπαγγελματικής ε, συμπεριφοράς και να αναλυφθεί η κατάλληλη δράση στην περίπτωση που γίνει αυτή η καταγγελία. Άρα ο ορισμός απαιτεί προσεκτική ανάλυση. Όπως ήδη ανέφερα, τα ζητήματα τα οποία καλύπτονται από το υφιστάμενο άρθρο 22α του κανονισμού θα πρέπει επίσης να συμπεριληφθούν δηλαδή περιπτώσεις στις οποίες ένας υπάλληλος λαμβάνει διαταγές στις οποίες αυτός ή αυτή θεωρεί παράτυπες ή ε, πιθανόν να οδηγήσουν σε σοβαρές δυσκολίες το να εστιάσουμε στην ευθύνη των θεσμικών οργάνων και της ε, διοίκησής τους στο να αναλάβουν αυτή η δράση νομίζω πως είναι το σωστό επί της αρχής. Και επίσης θα διορθώσει μια ανισορροπία η οποία υπάρχει σε φυστάμενες διατάξεις. Όπως εξέγησα, οι διατάξεις αυτές ε, επικεντρώνονται στο καθήκον καταγγελίας και στην αρνητική απέτηση μη αντικδίκηση, θα λέγαμε, των θεσμικών οργάνων ει βάρο των καταγγελόντων. Δεν ενθαρρύνουν την καταγγελία ω ένα μέσο ε, για να εκτελέσουν οι διοικούντες ε, της, ε, για να λάβουν διοικούντες ευθύνες τους. Υπάρχει εδώ πέρα βεβαίω μια λογική, καθώ ο καταγγέλων θεωρείται μια απειλή ή μια ενόχληση. Και πρόκειται για μια λανθασμένη προσέγγιση, γιατί έτσι γίνονται χειρότερα τα πράγματα. Η σωστή προσέγγιση είναι να βλέπουμε τι καταγγελίε ω μια ευκαιρία για να λάβουμε χρήσιμε πληροφορίε, να εξηγήσουμε τι πράξει αυτέ και να προχωρήσουμε σε διόρθωση, εάν αυτό απαιτείται. Όσον αφορά τον Όλαφ, η άποψή μου είναι πω ο νομοθέτη θα πρέπει να ορίσει σαφώ, με απλή γλώσσα, το πεδίο εφαρμογής της ε, αρμοδιότητας ερευνών του Όλαφ. Επίσης θα πρέπει να διασφαλιστεί πως ο κανονισμός περισσιακής κατάστασης και ο κανονισμός του Όλαφ ε, είναι συνεπής εδώ πέρα. Η άποψη μου λοιπόν είναι πως στόχος θα έπρεπε να είναι να, να βοηθήσει ο Όλαφ στην ηθική συμπεριφορά και να μην απαλλάξει τα θεσμικά όργανα από τις ευθύνες τους. Ο ρόλος τους να είναι ανακάλυψη περιπτώσεων απάτης, ε, διαφθοράς ε, κτλ. θα πρέπει να διαμορφωθεί αναλόγως. Είναι προφανές πως οι εσωτερικές έρευνες θα πρέπει να γίνονται από τον Όλαφ όταν αφορούν τη βασική του αρμοδιότητα, δηλαδή απάτη και διαφθορά. Δεν είναι όλες οι περιπτώσεις όμως κακής συμπεριφοράς απάτη και διαφθορά και θα πρέπει να μπορούν να κάνουν τις δικές τους διοικητικές έρευνες στα θεσμικά όργανα ε, όπου δει, όπως προβλέπει το άρθρο 86 του κανονισμού αυτή τη στιγμή. Το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο δεν προβλέπει αυτή τη στιγμή διαβούλευση μεταξύ όλαφ και θεσμικών οργάνων για το ποιο είναι σε καλύτερη θέση να ε, διεξάγει μια τέτοια έρευνα. Ούτε υπάρχει η δυνατότητα να ζητηθεί από τον Όλαφ τεχνική αρρωγή στο πλαίσιο μια εσωτερική έρευνα. Αυτά τα κενά θα πρέπει να αντιμετωπιστούν. Η πρόταση της Επιτροπής για τον οργανισμό του Όλαφ κινδυνεύει να κάνει τα πράγματα ακόμη χειρότερα, γιατί κατ' ουσίαν προβλέπει μια μονομερή απόφαση του Όλαφ για το εάν θα αναλάβει μια εσωτερική έρευνα ή όχι. Εάν αποφασίσει να κάνει κάτι τέτοιο, το εν λόγω θεσμικό όργανο δεν έχει την δυνατότητα να ξεκινήσει δική του έρευνα για τα ίδια γεγονότα. Και μάλιστα θα πρέπει να κλέσει και τυχόν έρευνες οι οποίες έχουν ήδη ξεκινήσει. Αυτό θα μπορούσε να έχει ω συνέπεια το θεσμικό όργανο να μην μπορεί να αναλάβει καμία πειθαρχική δράση μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα του Όλαφ. Καμιά φορά μπορεί αυτή να είναι η σωστή λύση. Αυτό θα ε, ισχύει παραδείγματο χάρη αν υπάρχει υποψία απάτης ή διαφθορά. Σε άλλες περιπτώσεις όμω, ίσω είναι γρηγορότερο και αποτελεσματικότερο να κάνει το ίδιο το θεσμικό όργανο μια διοικητική έρευνα, πιθανώ σε, περιπτώσεις, σε κάποιες περιπτώσεις με την τεχνική αρρωχή του Όλαφ. Πλην των περιπτώσεων που υπάρχει υποψία απάτης ή διαφθορά, δεν νομίζω πω μια μονομερής απόφαση του Όλαφ θα πρέπει να είναι ο κανόνα. Σε άλλες περιπτώσεις θα είναι καλύτερο να προβλεφθεί διαβούλευση και συμφωνία μεταξύ Όλαφ και θεσμικού οργάνου. Εάν δεν είναι δυνατή η συμφωνία θα πρέπει να υπερισχύσει η άποψη του Όλαφ μόνο εάν θεωρήσουμε πως υπάρχει προστασία των οικονομικών συμφερόντων της κοινότητας. Θα ήθελα να προσθέσω ένα τελευταίο θέμα όσον αφορά την πειθαρχική διαδικασία. Αφορά την κατάσταση που προβλέπει το άρθρο 25 στο παράρτημα 9 του Κανονισμού Υπηρεσιακής Κατάστασης. Δηλαδή, εκεί όπου, όπως αναφέρει, διώκεται ένας υπάλληλο για τις, δύο, για τις ίδιες αυτές πράξεις. Το άρθρο 25, λοιπόν, ξανά στα αγγλικά, προβλέπει πως μια οριστική απόφαση θα ληφθεί για πειθαρχικά ζητήματα μόνο κατόπιν οριστικής απόφασης από το δικαστήριο το οποίο κρίνει την υπόθεση. Τέλος, ο Στόχος εδώ πέρα βεβαίως είναι σαφής και αναμφισβήτητο, αλλά εγώ θεωρώ πως πρέπει να εξετάσουμε δύο ακόμα ζητήματα. Πρώτον, η αγγλική διατύπωση φαίνεται πως ε, εννοεί πως το άρθρο 25 ξεκινάει να ισχύει όταν φτάσει ενώπιον ενός δικαστηρίου μια υπόθεση και σταματάει να ισχύει όταν εκδοθεί απόφαση από το δικαστήριο. Άλλε όμω γλωσσικέ εκδοχέ φαίνεται πως υπονοούν πως ξεκινάει με την αρχή της έρευνας η ισχύ αυτής της διάταξης και τελειώνει όταν εξαντληθούν όλες οι δυνατότητες ε, έφεσης στην απόφαση αυτή. Να σας αναφέρω και το γαλλικό κείμενο για να το καταλάβετε. Όταν ο υπάλληλο αποτελεί αντικείμενο διώξεων για τα ίδια γεγονότα, η κατάστασή του διευθετείται μετά από την απόφαση της δικαστικής αρχής που θεωρείται ε, δεδομένη, γεγονό, τετελεσμένο γεγονός. Βεβαίως όλα εξαρτώνται από τη γλωσσική έκδοση. Το αγγλικό κείμενο μιλά για acts, για συμβάντα, ενώ ε, η γαλλική έκδοση μιλάει για fe, facts. Αυτά θα μπορούσαν να επιληθούν εάν επανασυντάξουμε την διάταξη μέσα στα πλαίσια των ε, πειθαρχικών διώξεων ή διαδικασιών και ενώπιον δικαστηρίου με βάση ποινική δίωξη. Εν κατακλείδη θα ήθελα να σας ε, σκιαγραφίσω μία ιδέα. Πρόκειται για μία προσπάθεια μια απαρχή προσπάθειας επίλυσης του ζητήματος και θα πρέπει να γίνει διαβούλευση πριν λάβει νομική ε, μορφή. Σας είπα πώς δημιουργήθηκε ο Όλαφ. Οι ίδιες συνθήκες δημιούργησαν και την έλλειψη εμπιστοσύνης στη, στα κοινοτικά θεσμικά όργανα. Θεωρώ ότι ο Όλαφ εξ αρχής είχε μεγάλο φόρτο ε, με βάση προσδοκίες που δεν μπορούσαν να πραγματοποιηθούν, ότι δηλαδή θα πρέπει να ανταποκριθεί σε όλα τα ζητήματα που μπορεί να θίξουν καταγγέλλοντες. Αυτό φαίνεται και από το άρθρο 22β σε σχέση με αποκάλυψη στοιχείων στο ελεγκτικό συνέδριο, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Κοινοβούλιο και στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή δεν ξέρουμε τι θα πρέπει να γίνει, πώς θα πρέπει να τύχουν σε αυτές οι πληροφορίες. Στην περίπτωση του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή θεωρούμε ότι πρόκειται για παράπονα. Αλλά δεν ξέρω πώς οι άλλοι φορείς αντιμετωπίζουν τις πληροφορίες που λαμβάνουν από καταγγέλλοντες. Εάν ορίσουμε σαφέστερα τις αρμοδιότητες του Όλαφ, ίσως θα ήταν χρήσιμο να γίνει πιο εμπεριστατωμένο το άρθρο 22β. Θα πρέπει δηλαδή να γίνεται διαβούλευση, να ανταλλάσσουμε πληροφορίες για τις διαδικασίες και να δούμε πώς έχουν οι χρηστές πρακτικές σε σχέση με την επαγγελματική δεοντολογία. Η Επιτροπή έχει ε, ορίσει ένα πρόγραμμα κατάρτισης για θέματα δεοντολογίας και ίσως θα πρέπει να λάβει θεσμικό χαρακτήρα. Θα ήμουν έτοιμος να σας βοηθήσω σε αυτή τη διαδικασία αν προβλεφθεί. Σας ευχαριστώ. Κύριε Δεμεσουλαβητά, τα χειροκροτήματα δείχνουν το ενδιαφέρον της Επιτροπής μας. Euh, πριν αρχίσει η συζήτηση θα ήθελα να δώσω το λόγο στο ε, κύριο Ζωάνο ε, Λουί που είναι ε, δικηγόρος και εξειδικεύεται σε αυτά τα θέματα. Σας ευχαριστώ. Κύριε Μεσολαβητά, χρησιμοποιήστε έναν όρο που είναι απολύτως εύστοχος κατά τη γνώμη μου και που συνοψίζει την αίσθηση και τις δυσκολίες τις οποίες αντιμετωπίζει ένας δικηγόρος όταν βρίσκεται ενώπιον της Όλαφ για να συνδράμει ένα υπάλληλο. Μιλήσατε για ασάφεια. Θα ήθελα να σας εξηγήσω τι σημαίνει τα πρώτα λεπτά μιας ακρόασης ενός προσώπου που ε, εμφανίζεται ενώπιον της Όλαφ για ανάκριση. Διαπιστώνει τη ταυτότητά του και του αναγυγνώσκουν τα δικαιώματά του. Και του λέγουν ότι έχουν το δικαίωμα να μην αυτοκατηγορηθεί. Σωστό είναι αυτό. Ως προς τη διαδικασία που συναντά κανείς σε όλα τα κράτη-μέλη. Στην ποινική δικαιοσύνη θα προχωρήσω ακόμα παραπέρα. Στα κράτη-μέλη ο κατηγορούμενος έχει μέχρι και το δικαίωμα να ψεύδεται απέναντι στο δικαστή του. Είναι ένα θεμελιώδης δικαίωμα. Μπορεί καμιά φορά αυτό να είναι θεμελιώδης, ε, ε, θεμελιώδης φάλμα της ε, υπεράσπισης. Και του διαβάζουν και άλλα δικαιώματα. Ότι έχει δικαίωμα να εκφραστεί σε όλες, σε οποιαδήποτε από τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά η έρευνα έχει πάντα μία γλώσσα που είναι τα αγγλικά ή τα γαλλικά. Με άλλα λόγια εξηγούν ξεκάθαρα στον ενδιαφερόμενο ότι αν έχουν την ανέδεια να θελήσουν να εκφραστούν στη γλώσσα τους, μαλτέζικα ή σλοβένικα για παράδειγμα, θα ήταν τεράστιο πρόβλημα που θα ενοχλήσει τους πάντες. Λυπάμαι πάρα πολύ, ακόμα και αν το λέει αυτό η κλήτευση και μόνο το γεγονός ότι αναφέρει ότι η έρευνα διεξάγεται στην εξή γλώσσα και εσείς έχετε το δικαίωμα να μιλήσετε άλλη γλώσσα. Γνωρίζουμε εξ αρχής ότι αυτό θα ε, συνδέεται με προβλήματα και δυσκολίες. Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα να ορίζεται η γλώσσα της διαδικασίας, αλλά ταυτόχρονα όταν αναφέρετε ότι έχετε δικαίωμα να ζητήσετε άλλη γλώσσα, είναι βεβαίως ασάφεια και προβληματικό. Και συνεχίζουμε τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις. Του λένε λοιπόν ότι δεν είναι υποχρεωμένος να αυτό κατηγορηθεί και να ε, καταθέσει εις βάρος του, αλλά του λένε προσοχή. Από τη σύσταση της Όλαφ και τις αποφάσεις που το διέπουν έχετε ε, την υποχρέωση να συνεργαστείτε πιστά με την Όλαφ και αυτό είναι ασφα... Ε, και αμφισημία και μάλιστα είναι θεμελιώδη παράληψη ή λάθος δικαίου και εκπορεύεται από την ίδια τη φύση του έργου της Όλαφ. Τι κάνει η Όλαφ. Διεξάγει μια διοικητική έρευνα. Για εσωτερική πάντα έρευνα πρόκειται ανάκριση, εξέταση του ε, προσωπικού. Βάσει ε, του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης, ο υπάλληλος, μόνιμος ή έκτακτος, ε, ε, οφείλει πίστη στο θεσμικό του όργανο. Θα πρέπει επίσης να σέβεται και την αξιοπρέπεια Κατά την άποψή μου λοιπόν, κάθε υπάλληλο και κάθε έκτακτος που ψεύδεται ε, κατά του θεσμικού οργάνου διαπράττει σοβαρότατο παράπτωμα διότι διαρριγνύει την απαραίτητη εμπιστοσύνη που θα πρέπει να ε, υπάρχει ανάμεσα στο θεσμικό όργανο και τα μέλη του προσωπικού. Και αυτή είναι ασάφεια και αμφισημία και είναι πάρα πολύ ενοχλητικό αυτό. Δηλαδή, μπορεί να έχουμε προετοιμάσει εμείς τον πελάτη μας, τον εντολέα μας, αλλά από τη στιγμή ε, που τους λέει ένας υπάλληλος του Όλαφ ότι δεν είστε υποχρεωμένοι να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις για να μην κατηγορήσετε τον εαυτό σας, αυτό ε, στην πραγματικότητα δεν ανταποκρίνεται στην ίδια τη ζωή. Γιατί λοιπόν υπάρχει αυτή η ασάφεια και η αφησιμία. Αυτή την εβδομάδα ήμουν στον Όλαφ σε μια τέτοια ακρόαση Και παρά τα όσα είπα στην Επιτροπή σας πριν από μία πενταετία, παρουσιάστηκε, συστήσαν μάλλον κάποιον ε, εκπρόσωπο ως δικαστή από κράτος μέλος. Αυτό το πράγμα είναι απαράδεκτο. Δεν έχω απέναντί μου δικαστή. Έχω υπάλληλο ή μόνιμο ή έκτακτο της Όλαφ και δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να δράσει ως εθνικός δικαστής. Δεν υπάρχει κανένα σατανικό στοιχείο εδώ. Αλλά νομίζω ότι αυτό που είναι εξωφρενικό είναι ότι τα μέλη του Όλαφ που κάνουν τις ε, ανακρίσεις δεν έχουν καταλάβει ότι όταν γίνονται μέλη του προσωπικού ενός θεσμικού οργάνου της Ένωσης δεν είναι πλέον δικαστές μπορεί απέναντι στις εθνικές τους αρχές να διατηρούν αυτή την ιδιότητα, αλλά όταν ε, είναι υπάλληλοι μόνιμοι έκτακτοι της Όλαφ, έχουν άλλη ιδιότητα που για μένα είναι ανώτερη και υπό την ιδιότητα αυτή διεξάγουν έρευνες και όταν παρουσιάζονται ως δικαστές εξαπατούν ε, τον υπάλληλο που ε, υφίσταται την ακρόαση αυτή τη ανανάκριση. Αυτό είναι πολύ μεγάλη αφησιμία, ασάφεια και δυσκολία για μένα ως δικηγόρο. Άλλη ασάφεια. Μας λέγουν ότι πρόκειται για διοικητική εξέταση. Στην πράξη όμως μπορεί να έχει ως συνέπεια τη στιγμή που ολοκληρώνεται τη διαβίβαση στις δικαστικές αρχές της χώρας και οι δικαστικές αρχές της χώρας μπορούν να αποφασίσουν κάλλιστα ότι θα κλείσουν ε, το θέμα και δεν θα ε, γίνει δικαστική έρευνα. Θα το στείλουν στο δικαστή που θα αποφανθεί επί της ουσίας βάσει ε, της έκθεσης του Όλαφ. Δεν είμαι πεπισμένος ότι αυτό είναι σύνομο, αλλά είναι άλλη ιστορία. Για μένα ως ε, Βέλγο θα πρέπει την έρευνα αυτή να την κάνει κάποιος αξιωματικός ε, της δικαστικής αστυνομίας στο Βέλγιο. Εν περιπτώσει, αυτό είναι σοβαρό θέμα, δεν ξέρουμε προς τα που ε, θα εξελιχθεί και πιστεύω ότι αυτά τα στοιχεία είναι πάρα πολύ σοβαρά διότι αμφισβητούν την ένομη ασφάλεια, την ασφάλεια δικαίου μάλλον που είναι εκ των όνων σε μια ευνομόμενη κοινωνία. Οπότε, εφόσον πρόκειται για διοικητική εξέταση και έρευνα, εκείνος που ερευνάται έχει ένα δικαίωμα, το οποίο δικαίωμα είναι η πρόσβαση στα στοιχεία, στα έγγραφα, τουλάχιστον τη στιγμή που κλείνει ο φάκελος. Αν είτε στη δικαιοσύνη θα έχει δικαίωμα ε, μετά το τέλος της έρευνας και πριν φτάσει στην ακροματική διαδικασία να δει τα έγγραφα. Εδώ δεν έχει καμία πρόσβαση ο ενδιαφερόμενος στο φάκελο του Όλαφ. Ουδέποτε. Τη μόνη στιγμή που θα έχει πρόσβαση στο φάκελο είναι εάν επαναπευθεί ε, στην εθνική του δικαιοσύνη ή στο e-doc που θα διαβιβάσει τι. Α, αυτό που είχε την ευγενή καλοσύνη να του στείλει η Όλαφ. Αλλά εγώ ως δικηγόρο δεν έχω καμία δυνατότητα να έχω πρόσβαση στο σύνολο του φακέλου, στο σύνολο των ε, ε, στοιχείων και των εγγράφων που χρησιμοποιεί ο Όλαφ. Και πολύ συχνά οι έρευνες είναι χιλιομετρικές, είναι τεράστιες. Δηλαδή και σέβομαι πάρα πολύ τους ερευνητές, αλλά ε, αν βάλουμε τα στοιχεία το ένα πάνω στο άλλο θα φτάσει στα 3-4 μέτρα ο φάκελος ύψος ε, χωρίς κανείς ποτέ να έχει πρόσβαση σε όλα αυτά τα έγγραφα. Οπότε εδώ πρόκειται πραγματικά για παραβίαση των δικαιωμάτων της υπεράσπισης και των βασικών αρχών, μεταξύ αυτών της αρχής ασφάλειας δικαίου. Και εκεί αυτόματα υπάρχει και ένα στοιχείο πάρα πολύ σοβαρό, που είναι η ίδια η έρευνα για τις διαδικασίες Όλαφ. Για ποιο λόγο αυτές οι έρευνες δεν ολοκληρώνονται ποτέ. Ε, πρώτος λόγος είναι ότι οι ερευνητές της Όλαφ δεν διαθέτουν τα απαραίτητα εκείνα μέσα που χρειάζονται για να φέρουν σε πέρας μια έρευνα με σωστό τρόπο. δεν έχει καθένας μία υπόθεση να χειρίζεται, αλλά 50.000, 100.000 κατακαιρματισμένα και ε, σκορπίζονται. Αυτό είναι πολύ <laughs> ωραίο για την οργάνωση του Όλαφ, αλλά είναι απαράδεκτο και αφόρητο για ένα ε, υπάλληλο έκτακτο ή μόνιμο που είναι αντικείμενο έρευνη. Και για μένα είναι απαράδεκτο κυρίω και αφόρητο για το θεσμικό όργανο που θα πρέπει να εργάζεται με κάποιον ε, εργαζόμενο που βρίσκεται σε μια κατάσταση αβεβαιότητας και που το μυαλό του είναι αλλού και όχι σε αυτά τα θέματα που χειρίζεται. Για ποιο λόγο ε, έχει τόσα προβλήματα Όλοφ, έχει σοβαρά προβλήματα, διότι όταν μια ανάκριση ή ακρόαση λαμβάνει χώρα, είναι δύο οι ανακριτές. Που συχνά εργάζονται σε μια γλώσσα που δεν είναι η μητρική τους και θα πρέπει να εξετάζουν ένα πρόσωπο. Οι απαντήσεις είναι συχνά πάρα πολύ μακροσκελείς, περίπλοκες και θα πρέπει να συνοψιστούν για να μπορέσουν να χρησιμοποιηθούν σε ένα πρακτικό συνεδρίασης. Οπότε χρειάζεται περίληψη σε μια γλώσσα που δεν είναι η μητρική, επαναλαμβάνω, του ανακριτού και αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολη υπόθεση. Και επιπλέον Καθώς οι ανακριτές του Όλαφ δεν έχουν ούτε βοηθό κανονικά ούτε γραμματέα για να κρατάει πρακτικά, να δακτυλογραφεί τη μαρτυρία, δεν θα πρέπει απλώς να ακούει, να παρατηρεί, να συνθέτει, αλλά να δακτυλογραφεί ε, ταυτόχρονα τις δηλώσεις. εμένα αυτό μου προκαλεί γέλια και κλάματα. Γιατί ως δικηγόρος εγώ είμαι επικουρικός της δικαιοσύνης και δεν μπορώ να δεχτώ ότι κάποιος δεν διεξάγει σωστά μια έρευνα. Και θα πρέπει κάποιο να χειρίζεται μια γλώσσα που δεν είναι η μητρική του, να δακτυλογραφεί χωρί ορθογραφικά λάθη. Ε, εκεί έχει το μυαλό του, εκεί επικεντρώνεται, οπότε δεν έχει τον απαραίτητο χρόνο για να κοιτάζει στα μάτια τον εξεταζόμενο για να πάει να του ε, αποσπάσει την αλήθεια από το βάθος των οφθαλμών του και του βλέμματός του δεν μπορεί να είναι απασχολημένο με άλλα θέματα που δεν είναι ζητήματα τη ανάκρισης, τη ακρόαση και τη εξέταση. Την αλήθεια τη βρίσκει κανείς και την αναζητεί στο βάθος του βλέμματος του ε, προσώπου και όχι στην οθόνη που γράφουμε τα πρακτικά εκείνη την ώρα. Και επανειλημμένα σας διαβεβαιώ ως δικηγόρος άκουα τις σφαίρες να με πλησιάζουν και να σφυρίζουν στα αυτιά μου με τον αέρα γιατί πραγματικά πλησιάζαμε, πλησιάζαμε, πλησιάζαμε και αρκούσε να ε, απλώσει κανείς το χέρι του για να πάρει το, το όριμο φρούτο. Στο layout περνούσαμε σε άλλη ερώτηση και είχε χαθεί η ανάκριση γιατί ακριβώς την κρίσιμη στιγμή δεν είχαν κάνει την ερώτηση που ε, ήταν απορρέουσα από την προηγούμενη απάντηση. Αλλά επειδή οι ε, ερωτήσεις ήταν έτοιμες εκ των προτέρων, δεν υπήρχε εκεί απάντηση, απέτυχε να βάγισε η διαδικασία της ανάκρισης εξέτασης και αυτό ήταν πάρα πολύ κακό, ολέφριο για τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης. Εγώ μπορεί να είμαι εκεί για να υπερασπίζομαι τους εντολείς μου και τους πελάτες μου, αλλά ο καλός εννοούμενος ρόλος ενός δικηγόρου όταν ε, ε συμπαρίσταται σε έναν πελάτη είναι να σέβονται τα δικαιώματα τη υπεράσπιση. Εμείς βοηθούμε τη δικαιοσύνη. Εμείς δεν έχουμε το δικαίωμα να δίνουμε μασημένη τροφή ε, στους πελάτες μας, να τους έχουμε μάθει ένα πείμα απ' έξω το οποίο να αναμασούν. Και λυπάμαι πάρα πολύ που να βάγει σε μια έρευνα, όχι επειδή είναι κακός ο ανακριτής, αλλά γιατί δεν έχει στη διάθεσή του τα μέσα που χρειάζεται για να κάνει σωστά τη δουλειά του. Συνέπεια όλων αυτών επίσης είναι ότι είναι ατέρμονες αυτές οι διαδικασίες και οι έρευνες. Οχτώ κροάσεις είχαμε σε μία και μόνο περίπτωση που διήρχησαν 55 ώρες συνολικά για ένα μέλος ε, της ε, μεσαίας διοίκησης. Και αυτό σημαίνει ότι ο εξεταστής είναι τελείως ακατάλληλος δεν ξέρει τι σημαίνει ο όρος ανάκριση ή εξέταση. Όταν πήρε το φάκελο, χρειάστηκε δύο χρόνια για να το μελετήσει. Αποκόμισε μια προσωπική ιδέα, ήταν μια υπόθεση επιδοτήσεων και θεώρησε ότι το έργο αυτό δεν έπρεπε να είχε χρηματοδοτηθεί, ενώ ο τμήματάρχης μου είπε, ξέρετε, εγώ αυτό το έργο ούτε καν δεν το είχα διαβάσει, γιατί ο δικός μου ρόλος είναι απλώς να βεβαιωθώ ότι οι επιρογνώμονες που έχουν επιφορτιστεί να γνωμοδοτήσουν για το έργο δίνουν τη γνωμοδότησή τους σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Συμπέρασμα αυτών των καθυστερήσεων. Πρώτον, αποβίασαν δύο άνθρωποι, εκ των οποίων ένα κλειδί που θα μπορούσε να είχε δώσει και ε, ε στοιχεία. Οπότε χάθηκε, έκλεισε η έρευνα αν είχε δράσει εγκαίρως, ε, επειδή όλα είχε ειδοποιηθεί πάρα πολύ νωρί για τα γεγονότα, θα μπορούσε να γίνει η ανάκριση και η εξέταση πάρα πολύ γρήγορα και να ολοκληρωθεί. Δεύτερη συνέπεια. Ήταν πολύ σημαντικές αυτές οι επιδοτήσεις ε, που χειριζόταν αυτό το τμήμα. Μετατέθηκε ο τμήματάρχης που πλέον σε άλλη υπηρεσία δεν χειρίζεται χρήματα. Αυτό είναι πραγματικά αξιοθρύνητο για την Ένωση. Ο άνθρωπος είναι ε, πάρα πολύ καλός υπάλληλο, ε, είναι θαυμάσιος στη θέση του, αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση έχασε ένα καλό υπάλληλο που είναι σε θέση να ε, χειρίζεται πολύ καλά αυτά τα οικονομικά θέματα και να τραβάει και κόκκινες γραμμές. Το 2004, πάω παρακάτω, είχε ανοίξει αυτή η έρευνα. Το 2008 άρχισα να εκνευρίζομαι, γιατί δεν είχε ολοκληρωθεί. διαβιβάσαμε στη συνέχεια, γιατί κατά σύμπτωση πρόκειται φυσικά για ανώνυμη επιστολή και θα το συζητήσουμε αυτό για το whistleblowing, την καταγγελία και τις ανώνυμες καταγγελίες σε λίγο. Nous avons... Λοιπόν, κατά σύμπτωση, εντελώ τυχαία, καταφέραμε να εντοπίσουμε, να ταυτοποιήσουμε τον συγγραφέα όχι το, της ανώνυμης επιστολής, αλλά εκείνο που είχε γράψει το φάκελο στο Γενικό Διευθυντή και διαβιβάζοντας εκείνος το φάκελο στο Γενικό Διευθυντή της Όλαφ είπε ότι δεν μπορώ καθόλου να αποκλείσω ότι πρόκειται για εσωτερικό ξεκαθάρισμα λογαριασμό, άρα είναι συγκοφαντική δυσφήμιση. Όλα αυτά τα διεκπαιρεώσαν. Ταυτοποίησαμε λοιπόν το συντάκτη, το συγγραφέα του φακέλου με γραφολογική εξέταση και πραγματογνωμοσύνη. 95,8% είναι η ασφάλεια ε, στη σύγκριση δύο δειγμάτων. Όλα θεώρησε ότι δεν χρειάζεται να ακούσει αυτόν τον άνθρωπο που είχαμε βρει ότι έγραψε το φάκελο. Τέσσερις μήνες αργότερα ρώτησα τι γίνεται με την έρευνα. Μου είπαν όλα καλά. Ε, συνεχίζει την πορεία της. Έχουμε φτάσει ήδη Απρίλιο 2009, πέντε χρόνια μετά τα γεγονότα. Μετά ψυχίστηκα ξανά αρχές του 2011 και μου είπαν λυπούμαστε πολύ αλλά εδώ και καιρό έχει τελειώσει η ερευνά σας και είναι στο αρχείο χωρίς συνέχεια. Α, μάλιστα. Αποφάσισε ο Όλαφ να θέσει όλα αυτά στο αρχείο αλλά ξέχασαν να ειδοποιήσουν τον ενδιαφερόμενο υπάλληλο. Α, ε, σιγά, λεπτομέρεια. Ανησυχούσε δύο χρόνια γονιούς ο άνθρωπος, δεν πειράζει. Δεν τρέχει τίποτα. Και μετά το διαβίβασαν στο ΙΝΤΟΚ που θεώρησαν ε, ότι δεν έπρεπε να αρχίσει έρευνα γιατί ήταν άδειο ο φάκελο. Μα δεν ελήφθη απόφαση από τον ΙΝΤΟΚ αφού δεν έγινε έρευνα. Αλλά θα μπορούσε να το ξαναστείλει στον Όλαφο όπως και έγινε και αποφάσισε να το βάλει στο αρχείο. Και περίεργο πράγμα, για δεύτερη φορά ξέχασαν να ειδοποιήσουν τον υπάλληλο και αυτό δεν έχει σημασία. Και εξ όσο γνωρίζουμε, ξέχασαν να ειδοποιήσουν και την αρμόδια γενική διεύθυνση ότι ήταν άδειο ο φάκελο. Αυτό που εμένα όμως με ενοχλεί περισσότερο από όλα αυτά είναι το εξή. Έστω, έστω, δέχομαι ότι υπήρξαν αξιόπινες πράξεις. Ποινικά κολάσιμες. Ε, επρόκειτο για ε, καταστάσεις που έγιναν το 2002-2003. Άρχισε ο φάκελος το 2004. Το 2011 ολοκληρώθηκε. Αν το είχαν αυτό διαβιβάσει στις ε, δικαστικές αρχές μιας χώρας, θα είχε παραγραφεί η υπόθεση. Αυτό είναι παράδεκτο στην Ένωση. Ε, λοιπόν, καταλαβαίνετε περί ποιας διάρκειας ομιλούμε υπάρχουν ε, προβλήματα και στις ικανότητες και στα μέσα, στην έλλειψη ικανότητων και έλλειψη μέσων που διαθέτουν οι ερευνητές και οι ανακριτές. Και κάτι άλλο που για μένα είναι δύσκολο να το δεχθώ. Όλαφ, σε μια υπόθεση που έλαβε τεράστια δημοσιότητα από τους ίδιους, γιατί Όλαφ έκανε συνέντευξη τύπου, σε ένα θέμα που υπήρχε υποψία για δίκτυο ε, δωροδοκία στο εσωτερικό των θεσμικών οργάνων. Ειδοποίησαν τους πάντες. Ξέραμε ακριβώς περίπου ποιες κατηγορίες προσώπων ήταν στο στόχαστρο. Η έρευνα άρχισε το 2004 και έκλεισε το 2011, ενώ μια εθνική έρευνα παράλληλα τρέχει ε, σε σχέση με τις εταιρείες και όχι τα πρόσωπα, έγιναν ακροάσεις σε ένα απίθανο, απίστευτο αριθμό προσώπων και πού κατέληξαν. Αθώωση για τους εννέα από τους 16 υπαλλήλου που ενέχονται και για τους υπόλοιπους 6 πραγματικά τι να σας πω. Dossier. Donc, διότι διαβιβάζεται ο φάκελος 7 χρόνια μετά την έναρξη στον IDOC και η επιστολή λέγει ότι παρόλο που δεν υπάρχει κανένας δόλος ή πρόθεση θεωρούμε ότι ορισμένα στοιχεία και ελλείψεις θα μπορούσαν να στοιχειοθετούνται εις βάρος. Ε, ναι, αν δεν υπάρχει πρόθεση, τι δουλειά έχει όλα σε αυτή την υπόθεση. Ακόμα περισσότερο να ε, βαρύνει την υπόθεση αυτή του ΙΝΤΟΚ. Και κάτι άλλο που είναι απαράδεκτο, κυρίως. Εδώ πρόκειται για υπαλλήλου που είναι άνθρωποι. Που έχουν μια πάρα πολύ μικρή ενημέρωση και πληροφόρηση. Είναι κατατρομοκρατημένοι, διότι δεν είχαν ποτέ δοσοληψίες με τη δικαιοσύνη. Και γιατί τόσες μακροσκελείς έρευνες. Το αποτέλεσμα είναι ότι καταστρέφονται αυτοί οι άνθρωποι αφενός και αφετέρου. Καταστρέφονται οι υπάλληλοι εκτός από άνθρωποι που δεν είναι σε θέση να εργάζονται όπως εργάζονταν στο παρελθόν, που έχουν χάσει όλες τους τις ελπίδες, τις ψευδεστήσεις τους, έχουν απογοητευτεί Και εγώ κάθε φορά που δέχομαι ένα πελάτη του λέω ε, θα πρέπει να πάρετε κάποια απόσταση από αυτή την κατάσταση. Αλλά η δέσμευσή τους, η προσήλωσή τους, η αφοσίωσή τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα είναι ποτέ ίδια. Και εγώ τους λέω να αποστασιοποιηθούν ακριβώς για να προστατευτούν από τους εαυτούς τους τους ίδιους. Σε σχέση με τον Όλαφ, θα πρέπει οπωσδήποτε να θεσπιστούν κανόνες παραγραφής για τις εσωτερικές έρευνες. Είναι απαράδεκτο να ανοίγουν διάφοροι φάκελοι για οτιδήποτε, να αρχίζουν έρευνες, όπως το είπατε και εσείς. Είναι απαράδεκτο η ε, Όλαφ να κάνει διοικητική έρευνα ε, που να μπαίνει στα χωράφια του ΙΝΤΟΚ. χωρίς να υπάρχει σαφής ε, απειλή για τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης. Και όταν τελειώνει η έρευνα της Όλαφ, έτσι κι αλλιώς ε, διαβιβάζεται στην EDOC, γιατί είναι υποχρεωμένη να κάνει τη διοικητική έρευνα ε, βάσει του παραρτήματος 9 για τις πειθαρχικές διαδικασίες. Σε ό,τι αφορά το E-DOC τώρα, θα πρέπει οπωσδήποτε να ε, τροποποιηθεί το παράρτημα 9 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης. Γιατί ποιο είναι για μένα το απαράδεκτο. Το πιο κατάφορο παράδειγμα ήταν οι γονότα που είχαν γίνει πριν από 22 χρόνια. Με κάποιες δηλώσεις, κάποια έγγραφα που είχαν κυκλοφορήσει πριν από 22 έτη. Το πρόβλημα που έχω ποιο είναι. Βεβαίως το δίκαιο δεν είναι κάτι το στατικό. Εξελίσσεται, όχι μόνο στα κείμενα, αλλά και στην εφαρμογή του και στην ερμηνεία του. Είναι σαφές ότι το ίδιο κείμενο συχνά, γιατί η κοινότητά μας είναι πάρα πολύ μεγάλη, με τρεις ε, βασικές έδρες. Λοιπόν, το ίδιο κείμενο δεν ερμηνεύεται κατά τον ίδιο τρόπο, αν πρόκειται για το Λουξεμβούργο, Στρασβούργο ή Βρυξέλλες. Σας ευχαριστώ την προσοχή στο γεγονός ότι, ε, για παράδειγμα, όταν άρχισε η μεταρρύθμιση, το Κοινοβούλιο είχε πολύ διαφορετική ανάγνωση για το πώς έπρεπε να τροποποιηθούν μερικές διατάξεις σχέση με την Κομισιόν ή άλλα θεσμικά όργανα. Λοιπόν, αυτά τα στοιχεία σιγά σιγά χάνονται και 22 χρόνια μετά δεν μπορεί κανείς να πει με τα Τι έγινε τότε που έγινε, εκεί που έγινε. Και από την άλλη ένα θέμα ασφάλειας δικαίου, όντω. Και είναι απολύτως απαραίτητο να οριστεί ένας κανόνας παραγραφής για οτιδήποτε ε, παράληψη ή συμπεριφορά που μπορεί κανείς να προσάψει σε ένα δημόσιο υπάλληλο. Αυτό υπάρχει παντού σε όλα τα κράτη-μέλη. Και είτε πρόκειται λοιπόν για ίντοκ, για όλαφ, για διοικητική ε, πειθαρχική ανάκριση, για όλα θα πρέπει να υπάρχει ένα νόημα για να προστατεύονται τα συμφέροντα των θεσμικών οργάνων και τα οικονομικά για την Όλαφ, ενώ για το EDOC είναι στα πλαίσια της επιθαρχικής διαδικασίας ε, τις περισσότερες φορές. Η πειθαρχική διαδικασία δεν έχει θεσπιστεί μόνο έτσι για την ευχαρίστηση που αισθάνεται κάποιο όταν τιμωρεί έναν υπάλληλο. Η καταδίκη από ένα εθνικό δικαστή, η φυλάκιση ή άλλη ποινή δεν είναι επειδή ευχαριστεί. Αλλά ο νόμος θα πρέπει να έχει ένα νόημα. Λοιπόν και η πειθαρχική κύρωση θα πρέπει να έχει νόημα. Δεν έχουμε το δικαίωμα στη δημοκρατία να τιμωρούμε για παραδειγματισμό. Θα πρέπει κάποιος να τιμωρείται ε, βάσει των πράξεών του και με τρόπο δίκαιο σε σχέση με αυτά που έκανε και σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο. Οπότε είναι προφανές ότι αυτή τη στιγμή έχει περάσει τόσος χρόνος από τις πράξεις αυτές και ε, ε, ο υπάλληλος είτε έχει μετανοήσει είτε έχει προχωρήσει και επιμείνει στη κατεύθυνση που είχε πάρει θα πρέπει να υπάρχουν κάποια όρια. και στις πιθανές πειθαρχικές κυρώσεις θα πρέπει να ενταχθούν δύο ακόμα στοιχεία που υπάρχουν στο εθνικό δίκαιο. Και αυτά είναι ε, η αναστολή, δηλαδή επιβάλλεται μία κύρωση αλλά αποφασίζεται να μην εφαρμοστεί σε περίπτωση που μέσα σε ένα λογισμένο διάστημα, ένα, δύο, τρία, πέντε χρόνια δεν υπάρξει υποτροπή, να μην εκτελεστεί. Ε, ή ε, σε αντίθετη περίπτωση να είναι πιο αυστηρή η ποινή. Και αν υπάρχουν ιδιαίτερες περιστάσεις, για να δούμε ε, γιατί κάποιος υπάλληλος δεν είχε τη σωστή συμπεριφορά. Σε περίπτωση λοιπόν που επιβληθεί μια πάρα πολύ βαριά ποινή, αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να ε, ανασταλεί αυτή, δηλαδή ε, τα γεγονότα είναι δεδομένα. Αυτό αναγνωρίζεται. Αλλά για λόγους σκοπιμότητας και τη στιγμή δεν επιβάλλεται η κύρωση. Αλλά αποφασίζεται ότι σε ένα χρονικό διάστημα που θα ορίσει η αρχή, αν δεν υπάρξει νέα καταδίκη, αν δεν υπάρξει νέο παράπτωμα, όλα αυτά χάνονται. Αν όμως υπάρξει και νέο παράπτωμα, ανοίγει ξανά ο φάκελος και κρίνεται το σύνολο των πραγματικών περιστατικών. Αυτό σημαίνει το εξής. Ε, σε πολλές περιπτώσεις καταλαβαίνει ο υπάλληλο πρώτον τη λάθος συμπεριφορά του, δεύτερον ότι είναι η τελευταία του ευκαιρία και τρίτον ότι αν ε, πέσει και σε άλλο παράπτωμα η ε, κύρωση θα είναι αμήλικτη και ακραία. Οπότε η ε, αναβολή ε, επιβολής ποινής και η αναστολή ε, είναι πραγματικά πολύ χρήσιμο γιατί δείχνει ότι το θεσμικό όργανο είναι διατεθειμένο να εμπιστευτεί τον υπάλληλο παρόλο που γνωρίζει ότι έχει υποπέσει σε ένα παράπτωμα αλλά του δίνει και άλλη μια ευκαιρία για να είναι δρυμύτερη την επόμενη φορά. Έτσι είναι οι διαδικασίες πιο ανθρώπινες για μένα, διαφυλάσσοντας πάντα όμως το συλλογικό συμφέρον και έχοντας και ελέγχοντας τη δυνατότητα να κάνουμε ε, ε, τον υπάλληλο να καταλάβει ότι εντάξει έγινε ε, μία φορά κάτι σοβαρό. Σε περίπτωση επανάληψης όμως θα πέσει ράβδος. Euh, Έχουμε 20 λεπτά στη διάθεσή μας. Προτείνω η συγγήτριά μας να ε, εκφράσει την άποψή της και θα το δούμε, θα δούμε και την άποψη της ε, διευθύντριας. Ευχαριστώ. Πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά να υπενθυμίσω πως είναι αυτή η πρώτη ακρόαση στο Κοινοβούλιο για το κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης ε, των υπαλλήλων, ένα θέμα που είναι ανοιχτό. Είχε γίνει, ξέρετε, παλιότερα και άλλη μια ακρόαση για τις ε, καταγγελίες και το θέμα είναι ακριβώς ποια είναι ε, η προσέγγιση τι γίνεται σε περίπτωση καταγγελίας και μετά από αυτά τα οποία άκουσα δεν ξέρω, εγώ θα πέτρεπα κάποιον από το να κάνει κάτι τέτοιο. Έχουμε λοιπόν ένα πρόβλημα γιατί έχουμε εξαιρετικές διατάξεις στο καταστατικό οι οποίες δεν αξίζουν τίποτα γιατί βλέπει ο καθένας το τι τον περιμένει εάν κάνει κάτι. Και υπάρχουν άνθρωποι στην αίθουσα που έκαναν κάτι τέτοιο και έχουν μια ιστορία πλέον που μας λυπεί και είναι τελείως αδιέξοδη. Ε, θα ήθελα επί τη ευκαιρία να ακούσω και την διευθύντρια του IDOC. Θα ήταν και αυτό ενδιαφέρον. Αλλά έχω και ένα ερώτημα σε σας, ε, Λουί. Ε, και σας, κύριε... Συνήγορε. Λέτε, ναι εντάξει, να υπάρξουν ε, οι διοικητικές ε, διαδικασίες. Αλλά ξέρετε στην ε, Κομισιόν απασχολείται μόνο το 40% του προσωπικού της κοινότητας. Με το υπόλοιπο 60% που δεν υπάρχει IDOC, τι γίνεται. Γιατί εδώ πέρα όλα φέχει κατ' ουσίαν μια μεγάλη διοργανική αρμοδιότητα. Οπότε πώς θα μπορούν οι καταγγέλλοντες να προστατευτούν όταν δεν υπάρχουν διαδικασίες. Κομισιόν από όσο ξέρω. Εντάξει, μπορεί να ισχύουν αυτέ οι παράγραφοι για όλα τα θεσμικά όργανα, αλλά το πώ εφαρμόζονται στα υπόλοιπα θεσμικά όργανα δεν είναι καθόλου γνωστό, γιατί δεν προβλέπεται τίποτα. Οπότε τι μα συμβουλεύετε να κάνουμε. Μπορεί να παραμείνει η παράγραφο για τι καταγγελίε ω έχει ή όχι. Μπορεί να παραμείνει και να λέμε πω ε, έχουμε αυτέ τι διαδικασίε και εξηγούμε το τι θα γίνεται με τι ε, καταγγελίε. Εάν όχι, θα πρέπει να α, αλλάξει και να ακούσουμε κάποιες απόψεις για το προς ποια κατεύθυνση θα πρέπει να πάει. Je vous propose c'est que chaque parlementaire s'exprime et qu'ensuite les questions soient, soient globalisées parce qu'il... Νομίζω ότι λαμβάνοντας υπόψη ότι έχουμε πολύ λίγο χρονικό διάστημα, δηλαδή 15 λεπτά, θα πρέπει να ολοκληρώσουμε τις εργασίες μας. Προτείνω λοιπόν να λάβει το λόγο ο συνάδελφός μας, Έπινγκς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, θα μιλήσω Ολλανδικά για να είμαι σαφέστερος. Εγώ εργάστηκα 7,5 χρόνια στην ε, Κομισιόν και τα τελευταία 2,5 χρόνια στο γραφείο το ιδιαίτερο του κυρίου Κάλλας, Επιτρόπου. με μεγάλη ευχαρίστηση εργάστηκα εκεί πέρα, αλλά είχα ένα ιδιαίτερο καθήκον εκεί πέρα. Ήταν το να προλάβω καταγγελίες από ανθρώπους. Γιατί η εμπειρία έχει δείξει, και συμφωνώ εδώ πέρα με την κυρία Γκρέσλε, πως οι καταγγέλλοντες ε, δεν είναι κάτι το οποίο εμφανίζεται ξαφνικά από τη μια μέρα στην άλλη. Δεν ξυπνάει κανείς ένα πρωί και του τη βαράει. Είναι μια σταδιακή διαδικασία. Είναι άνθρωποι με τις καλύτερες προθέσεις που υποτιμούν την δύναμη της γραφειοκρατίας του οργανισμού όπου εργάζονται και προσπαθούν μέσω της ιεραρχίας τους να κάνουν μια καταγγελία. Ίσως να μην πρόκειται βεβαίως πάντα για μια φοβερή απάτη. Είναι, μπορεί να είναι μικρά πράγματα, αλλά όπως σας είπα πρόκειται κατά κανόνα για αξιοπρεπείς ανθρώπους με τις καλύτερες προθέσεις. Αυτό το οποίο παρατηρούν λοιπόν γιατί σκέφτονται «Α, θα με προστατεύσουν όταν κάνω καταγγελία», είναι πως αποτελούν έναν ε, στόχο ακάλυπτο, γιατί πρέπει βεβαίως να το δηλώσουν στον ανώτερό τους ή πάνε στον ε, Όλαφ, όπου δεν ξέρουν πότε θα τελειώσει η υπόθεση. Υπάρχουν λοιπόν πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι θεωρούν πώς μπορούν να πέσουν στο καθεστώς αυτό του καταγγέλλοντος, αλλά μετά νομικά δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο. Τι γίνεται λοιπόν μετά. Α, παραμερίζονται. Εντάξει, δεν, ε, τους κλείνουν ε, σε κανένα δουλάπι, αλλά τους αγνοούν. Τους περιθωριοποιούν. Τους εξουδετερώνουν. Αν ήμασταν σε δικτατορία θα τους εκτελούσαν κιόλας. Αλλά βλέπετε πως το ίδιο μοτίβο επικρατεί. Και είχα... Ξέρετε πώς ξεκινάνε οι επαφές στις διάφορες γενικές διευθύνσεις με τους επιτρόπους λοιπά, για να πάνε, τους, να πάνε να βρουν τους ανθρώπους να πιούν ένα καφέ μαζί τους, να δουν τι γίνεται όντω και να προσπαθήσουν ίσως να λύσουν την υπόθεση για να μην φτάσουμε σε μια τέτοια κατάσταση, για να προστατεύσουν τελικά αυτούς τους ανθρώπους. Γιατί αν φτάσουμε σε αυτή την ε, υπόθεση και τελικά δεν καταλήξουμε σε μία ε, καταδίκη. Τι γη θα γίνει με αυτούς τους ανθρώπους. Κανείς μετά δεν θα τους θέλει. Θα πάνε από το ένα τμήμα στο άλλο, από τη μία γενική διεύθυνση στην άλλη. Κανείς δεν θα τους θέλει πουθενά γιατί είναι ο άνθρωπος που έκανε την καταγγελία και πάνε στο λεγόμενο Bureau de Passage. Κάθονται εκεί πέρα όλη τη μέρα και τους αφήνουν να σηκώνουν τα τηλέφωνα. Και αισθάνονται σε ένα πάρα πολύ μεγάλο οργανισμό τελικά πάρα πολύ μόνοι τους. Και καταραίει βεβαίως οποιαδήποτε ε, ιδέα είχαν για την Ευρώπη Ευρώπη κτλ. Οπότε, κυρία Γκρέσλε, για να είμαστε ε, δημιουργική. νομίζω πως θα μπορέσουμε να προστατεύσουμε πολύ περισσότερο αυτούς τους ανθρώπους, να δούμε τις ελλείψεις που υπάρχουν ε, στο καθεστώς αυτό, όταν μιλάμε για απάτη, Χωρίς αυτό βεβαίως να σημαίνει πως οποιαδήποτε κριτική ασκείται στην Κομισιόν είναι επίθεση ολόκληρο το σύστημα ή στο Γενικό Διευθυντή ή στην Ιεραρχία. Και θεωρώ άρα πως είναι πάρα πολύ σημαντικό ο κανονισμός να όσον αφορά την πρακτική του εφαρμογή. Μπορεί να έχουμε ένα πολύ ωραίο νομικό πλαίσιο, αλλά τελικά ε, οι άνθρωποι οι οποίοι θεωρούν πως κάτι είναι λάθος θα πρέπει να έχουν την δυνατότητα να το καταγγείλουν χωρίς να αποτελούν μετά ε, στόχο για τους υπόλοιπους. Αυτά και ευχαριστώ. Ο κύριος Έρενχάουζερ. Ευχαριστώ πολύ προσωπικά έχω δραστηριοποιηθεί και εγώ δύο φορές ως καταγγέλω. Την πρώτη φορά ήμουν φοιτητή και ήρθα αντιμέτωπο, με τη Στράμπακ που είναι ο δεύτερος κατασκευαστής στην Ευρώπη και είναι ύποπτη ότι ε, έχει δώσει μίζες στην Ουγγαρία ε, μέσω ενός κόμματος, ε, μιας εταιρείας μεσαζόντων ε, μας παρακολουθούσαν, μας έστειλαν ε, ιδιωτικούς detective, μας απείλησαν, προσπάθησαν και να μας δωροδοκίσουν, είχαν και συγκεκριμένη προσφορά και γενικά δεν ήταν σωστή η προστασία. Και το δεύτερο ήταν μόλις πρόσφατα, εγώ ίδιος έζησα το γεγονός ότι ο τότε ε, προϊστάμενος μου που τώρα είναι ύποπτος ότι είχε εξαιρέσει χρήματα ε, του κόμματος. Εκρεμούν και οι δύο υποθέσεις. Τι εννοώ, γιατί το λέω, γνωρίζω από προσωπική εμπειρία πόσο δύσκολο είναι όταν θέλει να καταπολεμήσει τη διαφθορά και τη δωροδοκία με τρόπο αποτελεσματικό θα πρέπει να υπάρχει μια σωστή προστασία των καταγγελόντων. Δεν υπάρχει αυτό σήμερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό που με κάνει αισιόδοξο είναι ε, η αναθεώρηση του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης είναι πραγματικά ε, μια πρώτη τάξεως και μοναδική ευθερία. Και το άρθρο 22α και το 22β θα πρέπει επιγόντως να ε, τροποποιηθούν, αλλιώς και τα επόμενα 20 χρόνια δεν θα έχουμε επαρκή προστασία. Τα τελευταία 10 χρόνια δεν ήταν πολύ μεγάλη η βοήθεια. Έχουν γίνει δύο μελέτες. Ε, η πιο πρόσφατη της Price Waterhouse Cooper την έχετε διαβάσει, την έχουμε συζητήσει εδώ στην Επιτροπή. Θα με ενδιαφέρει η απόψή σας. Και δεύτερη ερώτηση προς τον κύριο Διαμεσολαβητή. Έχετε κι εσείς περιπτώσεις τέτοιες καταγγελιών. Πόσες είναι αυτές και πώς τις αντιμετωπίζετε, τι κάνετε και ποιες είναι οι επιτυχίες σας σε αυτό το τομέα. Τρίτον, πάλι ερώτηση προς το διαμεσολαβητή. Έχουμε ενώπιόν μας ένα καταγγέλλοντο, τον κύριο Γκουίντο Στρακ. Γνωρίζετε την περίπτωσή του, την είχατε αντιμετωπίσει. Από ό,τι κατάλαβα εγώ, γεγονός είναι ότι οι αιτιάσει επί της ουσίας ή καταγγελίες δεν έχουν επί της ουσίας ε, γίνει αντικείμενο επεξεργασία σε κανένα θεσμικό όργανο. Μόνο τη διαδικασία σκέφτονται και θεωρείται τελευταία χρόνια του έχουν φερθεί σωστά. Ε, θέλω να ρωτήσω κάτι και τον κύριο Λουί. Ένα σημαντικό στοιχείο είναι όταν αποφασίσει ο Όλαφ να διακόψει μια τέτοια διαδικασία μετά από καταγγελία. Και τι γίνεται όταν ο καταγγέλων θεωρεί ότι είναι αδικία για τον ίδιο. Ποια είναι τα ένομα μέσα που διαθέτει, ε, τα ένδικα μέσα για να προχωρήσει, να προσφύγει κατά της Όλαφ και ποιες συνέπειες θα έχει Όλαφ και ο διευθυντής της όταν αποδειχθεί εκ των υστέρων ότι ε, ήταν σφάλμα η διακοπή της διαδικασίας. Ο κύριος Στράκ έχει υποβάλει εκτενή πρόταση για τροποποίηση του άρθρου 22α και 22β. Το, έχετε δει, ε, τη γνωρίζετε, θα με ενδιαφέρει η άποψή σας και η γνώμη σας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Υπάρχουν άλλες παρεμβάσεις. Εγώ εντάχει θα ήθελα να πω το εξής. Μιλάμε για άρθρα της υπηρεσιακής κατάστασης. φυσικά υπάρχουν ατέλειες, αλλά η υπηρεσιακή κατάσταση προσπαθεί να υπερασπιστεί τον υπάλληλο κατά τον ιεραρχικά ανώτερων, αλλά δεν τον υπερασπίζεται έναντι τρίτων. Δεν ξέρω δηλαδή κατά πόσο μπορούμε να επιλύσουμε διαφορές που κινούνται πέραν αυτού του πλαισίου, διότι μπορούμε να έχουμε να κάνουμε με μορφές οριζόντιας απάτης όπου εμπλέκονται πολλά θεσμικά όργανα. Αναρωτιέμαι λοιπόν κατά πόσο δεν θα πρέπει να γίνεται μία σύγκριση συγκριτική μελέτη στα κράτη-μέλη, γιατί στη χώρα μου υπάρχουν, υπάρχει το άρθρο 40 του ποινικού δικαίου που υποχρεώνει τον υπάλληλο να ε, αναφέρει τι συμβαίνει, τα συμβάντα. Και αυτό μπορούμε να το δούμε συγκριτικά και με το διεθνές ποινικό δίκαιο. Θα ήθελε η Διευθύντρια κάτι να ε, αναφέρει πριν δοθούν απαντήσεις γενικότερα σε σχέση με αυτά που ακούσατε. Δεν σας υποβάλαμε καμία ερώτηση συγκεκριμένα, απλώς μήπως, μήπως θέλετε να σχολιάσετε. Ερώτηση προς τη ευθύντρια. Ναι, ναι βεβαίως, δεν ήξερα πώς μπορούμε να κάνουμε ερωτήσεις. Βεβαίως θα με ενδιαφέρει. Η Κομισιόν έχει κάνει κάποιες πρώτες προτάσεις ήδη για την αλλαγή του καταστατικού. Για την προστασία των καταγγελόντων βλέπω δεν προβλέπεται κάποια αλλαγή. Θα με ενδιαφέρει να ακούσω ποια είναι η άποψη της Κομισιόν. Θεωρείτε πως ναι, χρειάζεται μεταρρύθμιση αυτού του άρθρου 22α και 22β. Θεωρείτε πως το χρειαζόμαστε τώρα και ότι είναι δυνατόν να γίνει στο πλαίσιο αυτής της ε, μεταρρύθμισης του καταστατικού και επίσης με ενδιαφέρει αυτό το οποίο ανέφερε και ο κύριος Διαμεσολαβητής. Υπάρχει και αυτή η μελέτη η οποία ήδη αναφέρθηκε στην Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Την έχετε διαβάσει, ποια είναι η άποψή σας για αυτήν. Ευχαριστώ. Thank you very much. Έχετε το λόγο. Καλό σας απόγευμα κυρίες και κύριοι. Λέγομαι Κάρεν Βίλιαμς και Είμαι διευθύντρια της IDOC, της Υπηρεσίας Ερευνών και Επιθαρχικών Εκυρώσεων, της Γενικής Διεύθυνσης Ανθρωπίνων Πόρων. Ε, χαίρομαι ιδιαίτερα που βρίσκομαι εδώ σήμερα το απόγευμα, γιατί θα ήθελα εντάχει να σας πω ορισμένα πράγματα, κατά πόσο τα άρθρα 21α και 21β θα πρέπει να αλλάξουν να αναμορφωθούν. Really need is... Συγχωρείτε, 22α και β πρέπει να αναμορφωθούν. Πρέπει να ανασυνταχθούν. Νομίζω ότι θα μπορούσαμε και θα επιβαλόταν να έχουμε ένα ενιαίο έγγραφο το οποίο να κοινοποιείται στο προσωπικό με όλες τις συνιστώσεις των στοιχείων καταγγελίας, δηλαδή γιατί γίνονται αυτές οι καταγγελίες. Μιλάμε για θέματα απάτης και διαφόρων όταν πρόκειται για σοβαρές περιπτώσεις. Εδώ δεν συμπεριλαμβάνονται τα πάντα. Και αυτό που έχει σημασία είναι να δούμε ποιοι διαδραματίζουν ποιο ρόλο, πώς μπορούν να προστατευτούν οι καταγγέλλοντες αποτελεσματικά και όλα αυτά θα πρέπει να εξηγούνται σε ένα έγγραφο το οποίο να είναι προσιτό σε όλους τους υπαλλήλους για να ξέρουν πώς έχει κατάσταση πιο ολοκληρωμένα. Ε, αυτές οι μορφές καταγγελίας είναι ένα από τα στοιχεία του οπλοστασίου για να δούμε κατά πόσο υπάρχουν παρατυπίες. Οι καταγγελίες παραπτωμάτων λοιπόν υπάρχουν για περιπτώσεις απάτης και διαφθοράς και υπάρχουν και άλλοι κανόνες για άλλες καταστάσεις ή συμβάντα. Θα πρέπει να δούμε πόσα όλα αυτά εντάσσονται και συνδέονται και ποιοι είναι οι μηχανισμοί και τα ε, στοιχεία κατεύθυνσης για το προσωπικό που θέλει να κοινοποιήσει κάτι, να κάνει μια καταγγελία, πού πρέπει να την υποβάλει την καταγγελία. Όλα αυτά θα πρέπει να επεξηγούνται λεπτομερώς. Ως προς τη μελέτη, διαβάσαμε τη μελέτη και θα ήθελα να ευχαριστήσω την Επιτροπή για η Επιτροπή Ποιοι ανέθεσε, μάλλον ζήτησε αυτή την έρευνα. Η House Coopers ε, διενέργησε αυτή την έρευνα. Υπάρχουν ορισμένες χρήσιμες υποδείξεις σε αυτή τη μελέτη που θεωρούμε και στοιχεία που μπορούμε να εντάξουμε στα πλαίσια αυτής της ανακοίνωσης. Γιατί Εν υπάρχει ένα νέο έγγραφο το οποίο ενημερώνει, επικαιροποιεί και συντάσσει όλα αυτά τα στοιχεία. Αυτό καθεαυτό θα επιτρέψει στο προσωπικό να γνωρίζει ότι αυτή η πλευρά της καταγγελίας είναι ένα αναπόσπαστο στοιχείο για την ίχνηλάτηση της διαφθοράς και της απάτης. κάτι το οποίο δέχεται η Επιτροπή και προωθεί μάλιστα, έτσι ώστε να προστατεύεται και ο καταγγέλων κατά το δυνατόν. και να ορίσουμε πότε μπορεί κάποιος να θεωρηθεί καταγγέλων και πότε όχι. Η κατάσταση για την Όλαφ είναι ίσως πιο σαφής, αλλά θα πρέπει να αποσαφινιστεί περαιτέρω. Ως προσορισμένα ε, στοιχεία που ανέφερε ο Ευρωπαίος ε, Διαμεσολαβητής και ο Μέτρ, σε σχέση με τον Διαμεσολαβητή θεωρώ ότι το θέμα ε, αυτής της προσέγγισης και οριοθέτησης έχει μεγάλη σημασία για να ορίσουμε κανόνες δεοντολογίας πρωτίστως μέσα στα πλαίσια της ανάληψης καθηκόντων από ε, προσωπικό ιεραρχικά ανώτερο. Στα πλαίσια της IDOC, και εγώ ασχολήθηκα με αυτό το θέμα προσωπικά, και αυτό που έχει σημασία είναι να δούμε πώς πιο αποτελεσματικά μπορούμε να μιλάμε στο προσωπικό, να γνωστοποιήσουμε την εργασία της ε, IDOC, της υπηρεσίας μου, μέσα στα πλαίσια του πειθαρχικού και να γνωρίζουν ότι φέρουν άμεση ευθύνη και για το προσωπικό τους, ιεραρχικά ε, ανώτεροι, και ότι φέρουν μεγάλη ευθύνη και στο πλαίσιο αυτό των καταγγελιών. Σε σχέση με την Όλαφ, καθε αυτή, γίνεται λόγος για μεταρρύθμιση του κανονισμού της Όλαφ. Νομίζω ότι το συζητήσατε σήμερα το πρωί. Αυτός ο κανονισμός σχετίζεται με τα χρηματοοικονομικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή είναι και η νομική βάση που διέπει τον κανονισμό. Υπάρχει επιμερισμός καθηκόντων μεταξύ Όλαφ και ΆΙΔΟΚ για τη διενέργεια ερευνών. Τα ζητήματα αυτά τα συζητάμε με την Όλαφ Έχουμε ένα ε, υπόμνημα συνεννόησης, ένα μνημόνιο συνεννόησης και καταβάλουμε κάθε προσπάθεια έτσι ώστε η σωστή υπηρεσία να διαχειριστεί την κάθε υπόθεση. Βεβαίως ε, μπορούμε να καταφέρουμε πολύ περισσότερα και πρέπει να υπενθυμίσω ότι ένας από τους βασικούς στόχους της μεταρρύθμισης αυτού του κανονισμού είναι ο εξής. Θα πρέπει να ορίσει να φτάσει μια καλύτερη ιεράρχηση της Όλαφ μέσα στα πλαίσια της ανάληψης ερευνών και αυτό το δεχόμαστε και το υποστηρίζουμε. Και γι' αυτό προσβλέπουμε σε αυτό τον αναθεωρημένο, τροποποιημένο κανονισμό ε, κατανοώ την κατάσταση του διαμεσολαβητή, διότι προσπαθεί να κατανοήσει το ρόλο της Όλαφ σε μη οικονομικά, χρηματοοικονομικά ζητήματα. Γιατί δηλαδή η Όλαφ πρέπει να διαχειρίζεται αυτές τις υποθέσεις. Και πρέπει κανείς να καταβάλει ιδιαίτερη προσπάθεια για να διασαφηνίσει ε, πού θα προέρχεται αυτός ο ρόλος. Εσείς βεβαίως κάνατε την έρευνά σας και είπατε ακριβώς ότι βασιζόσαστε σε αυτή τη διαθεσμική συμφωνία και όχι τον κανονισμό της Όλαφ καθεαυτό. Αυτό δεν προβλέπεται στο τρέχον πακέτο της μεταρρύθμισης, αλλά είναι ένα θέμα μεγάλου ενδιαφέροντος για το μέλλον και ίσως αυτό μπορούμε να το λάβουμε υπόψη για τους μελλοντικούς μας χειρισμούς. Ως προς τις προθεσμίες και την πρόσβαση στα αρχεία, ο Μέτρ Λουί μας εξέφρασε τις ανησυχίες του για, το, για τις υποθέσεις αυτές που είναι ιδιαίτερα σχηνοτενείς μέχρι ότου ολοκληρωθούν. Εγώ δεν μπορώ να μιλήσω εξ ονόματος της Όλαφ. Ο νέος κανονισμός όμως θα προσπαθήσει να υπάρχει μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα σε αυτό το τομέα. Εμείς ως IDOC έχουμε καταβάλει μεγάλες προσπάθειες για να μειώσουμε το χρονοδιάγραμμα των δικών μας ερευνών. Έχουμε καταβάλει υπεράνθρωπες προσπάθειες από το 2009 και έχουμε αυτούς τους ρυθμούς ακόμα. Αν δείτε την ετήσια έκθεση βλέπετε ο μέσος όρος διάρκειας της έρευνας είναι 6 μήνες. Και για πειθαρχικές διώξεις ένας χρόνος με 14 μήνες είναι το ανώτατο όριο. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη αυτές τις παραμέτρους για να είμαστε όσο πιο αποτελεσματικοί μπορούμε. Και ως προς το δικαίωμα υπεράσπισης των προσώπων μας ενδιαφέρει όλος ιδιαίτερος. Μέσα στα πλαίσια της πειθαρχικής δίωξης γίνεται ακρόαση του ενδιαφερομένου πολλές φορές πριν ληφθεί η απόφαση και στα πλαίσια αυτής της διαδικασίας υπάρχουν, δίνονται πολλές ευκαιρίες μάλλον στον ενδιαφερόμενο να εκφραστεί πριν ληφθεί η απόφαση από την αρμόδια αρχή για οποιαδήποτε πτυχή αυτής της υπόθεσης. Ως προς αυτό το φάσμα μέσων που έχουμε στη διάθεσή μας. Υπάρχει ένα ευρύ φάσμα κυρώσεων από τις οποίες μπορεί να επιλέξει κανείς και άρα η αρμόδια επί των διορισμών αρχή λαμβάνει υπόψη όλες τις παραμέτρους, δηλαδή το ε, πόσο έχει διαρκέσει αυτή η υπόθεση, αν πρόκειται για μια παλαιά υπόθεση, δηλαδή που έχει αρχίσει πολύ καιρό πριν. Όλα αυτά λαμβάνονται υπόψη στη λήψη απόφασης, διάρκεια της υπόθεσης και ούτω καθεξής. Ως προς θέματα χρόνου, έχει μεγάλη σημασία να λάβουμε υπόψη το, στη συνολική διάρκεια της υπόθεσης. και θα πρέπει να ερμηνεύουμε κατά τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο τις διατάξεις που ήδη έχουμε στη διάθεσή μας. Γι' αυτό υποστηρίζουμε αυτά που είπε ο Δία Μεσολαβητής σε σχέση με την ερμηνεία του άρθρου 25 της ε, υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων. Θα θέλαμε να ερμηνεύεται αυτή η διάταξη κατά τρόπον ώστε να μπορέσουμε να, έχουμε, να λάβουμε τις σωστές πειθαρχικές αποφάσεις, διότι όταν καθυστερεί η δικαιοσύνη δεν αποδίδεται στο τέλος. Έχει εκπνεύσει ο χρόνο της συνεδρίασης. Προτείνω να συνεχίσουμε στα αγγλικά, εκτός αν έχουμε ε, μια μικρή περίοδο χάριτος. Μας εκχωρούν οι διερμηνείς. Λίγη ώρα. Εντάξει. Να κλείσουμε λοιπόν δύο λεπτά απάντηση για κάθε ε, εισηγητή μας και η εισηγήτρια επίσης σε δύο λεπτά θα συνοψίσει την αίσθηση της. Ε, Ευχαριστώ. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομος, διότι μιλήσατε για την προστασία των καταγγελόντων. Θα πρέπει να μιλήσουμε γενικότερα για προστασία των whistleblowers. Να σας δώσω ένα παράδειγμα για το τι συμβαίνει σε ένα περιφερειακό θεσμικό όργανο και όχι ε, κεντρικό ε, της Ένωσης. Πάντως η Όλαφ έχει αρμοδιότητα εκεί. Κάποιος με μεγάλες επιφυλάξεις, γιατί πρόκειται για τον άμεσα προϊστάμενό του, δήλωσε στην ιεραρχία του κάποιες υποψίες για τα σταλίες παραπτώματα μέχρι και απάτη υπεξαίρεσης χρημάτων του αμέσως προϊσταμένου. Η αρμόδια αρχή του έδωσε την προστασία ε, του whistleblower, αλλά του είπε με την ιδιότητά σου αυτή δεν έχεις δικαίωμα να κάνεις η αδίποτε δήλωση. για τα γεγονότα για τα οποία καλύπτεσαι. Όταν λοιπόν έγινε εσωτερική έρευνα, δεν μπόρεσε ο ενδιαφερόμενος να μιλήσει. Και δεν μπόρεσε καν να δηλώσει ότι εκείνος είχε ενημερώσει τη διοίκηση για τις υποψίες του. Μη έχοντα αυτά τα στοιχεία, η διοίκηση το, τα διαβίβασε όλα αυτά στην Όλαφ που τον ε, άκουσε ως ε, μάρτυρα. Αλλά ο διευθυντής που του έδωσε αυτή την προστασία εντό εισαγωγικών, του είχε πει ότι δεν είχε το δικαίωμα να μιλήσει ακριβώς επειδή ήταν στο σύστημα προστασίας. Οπότε στα πρακτικά του Όλαφ, τρεις φορές δήλωσε ότι δεν μπορώ στο παρόν στάδιο της διαδικασίας να μιλήσω. Λογικά λοιπόν ο Όλαφ είπε, ακούστε, εγώ σας ακούω ως ενδιαφερόμενο μέρος. Και του είπαν και πάλι, όμως θα χάσετε την προστασία σας αν μιλήσετε. Με ρώτησε και του είπα, λυπάμαι πάρα πολύ, αλλά δεν μπορώ να δεχτώ να χάσει την προστασία του επειδή απαντάει στις ερωτήσεις σας. Πάρα πολύ γρήγορα. Το εκτελεστικό συμβούλιο αυτού του θεσμικού οργάνου, μη όντας ενήμερο για την κατάσταση αυτή, εξέτασε τη δυνατότητα να τον θέσει σε διαθεσιμότητα αποφάσισε προς το παρόν να μην το πράξει, αλλά του αφαίρεσε τη δυνατότητα υπογραφής Δηλαδή γνωρίζει όλο το θεσμικό όργανο ότι υπάρχουν σοβαρές περιστάσεις που δικαιολογούν να του αφαιρθεί η δυνατότητα υπογραφής. Αν αυτή είναι η προστασία του whistleblower, πολλοί ε, αμφιβάλλουν και εγώ έχω ενοχληθεί. Για μένα ποιο είναι το πρόβλημα, πάρα πολύ σύντομα θα πρέπει να προστατεύουμε εκείνο που καταγγέλει και δίνει πληροφορίες. Αλλά θα πρέπει επίσης να προστατεύουμε και τον κατηγορούμενο ε, προκειμένο Γιατί έχουμε πραγματικά καταστροφές, ε, φρικτές περιπτώσεις, γιατί είναι ξεκαθάρισμα λογαριασμών. Υφίστανται κάποιοι βαρύτατες κατηγορίες αποκλειστικά και μόνο διότι είχαν την ανέδεια να απαιτήσουν το προσωπικό που είναι υφιστάμενό τους να εργάζεται. Και ε, έγιναν καταγγελίες και μηνύσεις ε, για παρενόχληση και άλλα τιμά. Ε, δύο, υπόψεις, δύο υποθέσεις τέτοιες έχω υπόψη μου. Αυτό είναι σκέτη καταστροφή. Θα πρέπει να είναι σαφείς οι κανόνες. Για να απαντήσω λοιπόν στην ερώτησή σας είναι το άρθρο 22 ε, και 22α και θεωρούμε ότι, εγώ θεωρώ ότι το πλαίσιο είναι επαρκές για να δίδονται όλες οι ε, διευκρινήσεις όπως είπατε κυρία Διευθύντρια. Ας μην ξεχάσουμε επίσης το άρθρο 24 που επιβάλλει σε κάθε θεσμικό όργανο να προστατεύει ένα μέλος του προσωπικού από επιθέσεις που μπορεί να προέρχονται και έξωθεν. Υπάρχουν νομικέ βάσει, αλλά θα πρέπει να εφαρμόζονται στην πράξη, να τίθενται σε ισχύ και να προστατεύουν κάθε υπάλληλο. Και οι διαδικασίε αυτέ είναι ουσιώδει για την Ένωση. Ευχαριστώ, κύριο Διαμεσολαβητή, παρακαλώ. Um, σε δύο λεπτά και βεβαίω είναι αδύνατο να, να απαντήσω τι ερωτήσει. να προσπαθήσω τηλεγραφικά. Εγώ βλέπω μία σχέση μεταξύ των παρατηρήσεων του κύριου Έπιν και της κυρίας Βίλιαμς. Υπό την έννοια ότι επικροτώ τον κύριο Έπιν, που προσπάθησε βεβαίως να πει πως πρέπει να τεθεί το ζήτημα αυτό σε ένα ευρύτερο πλαίσιο και να μην υπάρχει καν η ανάγκη να κάνει κανείς την ε, καταγγελία. Για να μην έχουμε το όλα ή τίποτα δηλαδή. Οπότε πρέπει να υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη ευελιξία. Και καταλαβαίνω πως και η κυρία Williams είπε κάτι ανάλογο. καθώς είπε πως αυτό πρέπει να εξηγηθεί. Αυτή τη στιγμή εξηγούμε. Ε, ήδη υπάρχει μια κατεύθυνση για τις διάφορες φάσεις τις οποίες μπορεί να εξηγηθεί και να αποφορτιστεί και να επιληθεί μια ε, κατάσταση. Οπότε έτσι μπαίνει σε ένα πλαίσιο η καταγγελία που είναι ένα σημαντικό μέσο αλλά πρέπει νομίζω καλύτερα να ε, εξηγηθεί. Και τα άρθρα αυτά τα εφιστάμενα δεν το κάνουν και αυτό το λέω σαφώς. Δεύτερον, να πω στον κύριο Έρνχάουζερ ε, μου πήραν και εμένα συνέντευξη για τη μελέτη, είδα και εγώ τη μελέτη, συμφωνώ με την κυρία Williams, είναι περιγραφική, έχει βεβαίως κάποιες χρήσιμες ιδέες που μπορούν να υιοθετηθούν. Πράγματι είχα περιπτώσεις καταγγελιών γύρω στις 10-11. Δυστυχώς ε, είναι πολύ, πολλές εμπιστευτικές περιπτώσεις, οπότε δεσμεύομαι και δεν μπορώ παρά να σας πω μόνο πως είχα γύρω στις 10 τέτοιες περιπτώσεις. Γι' αυτό το οποίο είπε ο κ. Στρακ, κύριε Ρενχάουζερ, πράγματι πρόκειται για μια πολύ λυπηρή υπόθεση η οποία κατέληξε σε πλήρη διακοπή επικοινωνιών μεταξύ του καταγγέλλοντος και της ε, Κομισιόν και δεν μπόρεσα να διαμεσολαβήσω και εξέφρασα μόνο την μεγάλη μου απογοήτευση για την κατάσταση αυτή. Σαφώς δεν είναι η ιδανική κατάσταση. Ήταν λυπηρόν και για τον κύριο Στράκ και για την Κομισιόν το πώς εξελίχθηκε αυτή η υπόθεση. σταματήσω εδώ πέρα. Θέλω να ευχαριστήσω την κυρία Γουλιαμς για να πω πως συμμερίζομαι και εγώ τις ανησυχίες της και ελπίζω πως θα επανεξεταστεί η αποστολή του Όλαφ και να ξεκαθαρίσει. Δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμα και νομίζω που συμφωνεί εδώ πέρα και ο κ. Κέσλεφ. Είναι και η συγγήτριά μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Όσοι συμμετείχαν έχουμε μια παροιμία στα γερμανικά η οποία λέει όταν δεν ξέρεις να κάνεις κάνει μια επιτροπή. Ε, και εμείς εδώ πέρα βλέπετε πως έχουμε μια επιτροπή. Ο κύριος Λουίς μας είπε πως ε, τα πράγματα επαρκούν, ε, αρκεί να εφαρμοστούν. Ο κύριος Διαμεσολαβητής μας είπε πως οι κανόνες δεν επαρκούν. Ίσως και οι δύο να έχουν κάποιο δίκαιο και η επιτροπή αυτή, αν θέλετε, που ανέφερα, θα έπρεπε να βρει το τι θα κάνουμε. Έχουμε μια μοναδική κατάσταση, μια ευκαιρία να προχωρήσουν τα πράγματα, αλλά θα πρέπει να καταλήξουμε κάποτε κάπου και η ακρόαση έδειξε πως έχουμε πάρα πολλά στοιχεία. Ξεκινάει από τον Όλαφ, υπάρχει και το Άιντοκ στη μέση και εγώ θα ήθελα η Κομισιόν να είχε το θάρρος να προτείνει κάτι. Δυστυχώς στην πρόταση αυτή δεν υπάρχει τίποτα, οπότε φοβάμαι πως θα πρέπει να εργαστούμε εμείς με τα πενιχρά μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας. Αλλά ε, έστω και με κάποια non-paper η κυρία Williams μπορεί να μας κάνει κάποιες ε, προτάσεις δικιά της δουλειά θα ήταν, αλλά βεβαίως ε, ξέρετε πως ε, επειδή ε, έληφθη η απόφαση να μην γίνουν μεγάλες αλλαγές, καταλήξαμε να έχουμε μόνο τις ψυχές του προπολογισμού στην αναθεώρηση του καταστατικού και αυτό δεν το θεωρώ πάρα πολύ σωστό η έκκλησή μου προς την Κομισιόν είναι να έχει το θάρρος να λύσει τα προβλήματα που υπάρχουν εδώ και πάρα πολλά χρόνια στην, στον κανονισμό υπηρεσιακής ε, κατάστασης. Οπότε σας ευχαριστώ, ευχαριστώ και την Γενική Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων και όλους τους συμμετέχοντες. Ευχαριστώ κύριε Δημασολαβητά, κύριε Λουί Ίγκε. Κύριε Γουίλιαμς, ε, η πάλα είναι στο γήπεδό σας λίγο, το καταλάβατε. Ευχαριστώ πάρα πολύ και τους διερμηνείς, γιατί εμείς τέμε, ε, αργήσαμε να αρχίσουμε. Ευχαριστώ πολύ. Πολύ εντυπωσιακή αυτή η συζήτηση και πάρα πολύ χρήσιμη για τους υπαλλήλους μας που πρέπει να προστατεύονται. Ευχαριστώ πολύ.